Καλημέρα συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ακρόαση. Συμπροεδρεύουμε και οι δύο, κύριε Μασίτα και εγώ. Κοινή ακρόαση επιτροπών ΛΥΜΠΕ και γυναικών. θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των προσκεκλημένων μας όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Ένα ε, εξαιρετικά σημαντικό νομοθέτημα και για τις δύο επιτροπές μας και φυσικά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία έθεσε σε εφαρμογή έναν μηχανισμό για την ε, αμοιβαία αναγνώριση σε ποινικά ζητήματα και ε, έπρεπε να μεταφερθεί ε, το νομοθέτημα αυτό ε, στην Εθνική Νομοθεσία των Κρατών Μαλών έως τον Ιανουάριο του 2015. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια και ακόμη υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της έντολης προστασίας. Μέχρι στιγμής μόνο 7 έχουν, ε, τέτοιες εντολές έχουν εκδοθεί, κάτι που μας ανησυχεί πολύ. Και βεβαίως τα μέλη αναμένεται να μιλήσουν για αυτό το θέμα, όπως και εγώ και η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών. Η μεγάλη ποικιλομορφία στα νομοθετήματα, στο νομοθετικό πλαίσιο, η περιπλοκότητα των μέσων αυτών, αλλά και η ελπή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι κάποια από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από την αξιολόγηση του EPRS, που επίσης θα ε, παρουσιαστεί σήμερα όσον αφορά αυτή την περιορισμένη χρήση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων και ε, θα μας βοηθήσει στην σύνταξη μιας έκθεσης που πρόκειται να συντάξουμε ε, βάσει του άρθρου 55 στο προσεχές διάστημα. Εισαγωγικά αυτά ήθελα να πω και να δώσω τώρα το λόγο στην, ε, στην Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράες. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω όλα τα μέλη των δύο επιτροπών. Αυτή, αυτές οι κοινέ συνεδριάσεις πραγματικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολύ χρήσιμες λόγω των πολλών κοινών θεμάτων που μας απασχολούν ως επιτροπές αλλά και τις πολύ καλές σχέσεις εργασίας που έχουμε πλέον ε, δημιουργήσει μεταξύ των δύο επιτροπών. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας λοιπόν ήταν ένα λογικό βήμα ε, στον τομέα των ε, μηχανισμών προστασίας που μπορούν να εκδίδουν τα κράτη-μέλη. Στη, βάση της αξιολόγησης ε, που προηγήθηκε της οδηγίας 100.000 γυναίκες έχουν τύχη προστασίας από εντολή προστασίας. Ε, χρίζουν προστασίας. Γι' αυτό και οι γυναίκες αυτές κατά κύριο λόγο θα ήταν ε, οι δικαιούχοι αυτές, αυτής της εντολής προστασίας κατά την ε, διαμονή τους ή την μετακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ωστόσο, παρά την, τις μεγάλες ανάγκες, μόλις 7 τέτοιες ευρωπαϊκές εντολές προστασίας έχουν εκδοθεί. Είναι πραγματικά σοκαριστικός αυτός ο αριθμός και ελπίζω ότι η ακρόαση θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει και στη σύνταξη της κοινή έκθεσης ε, που προετοιμάζουν οι δύο επιτροπές μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής αυτής της εντολής οι, οι πρώτοι ομιλητές που θα λάβουν το λόγο είναι οι δύο συνεισηγητές μας των δύο επιτροπών. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, κύριο Ράιοπος. Έχετε πέντε λεπτά παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. And good... Κύριε ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι και εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή και η σημερινή ακρόαση είναι πολύ σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που πραγματικά αποτελεί ντροπή που δεν έχουμε καταφέρει να το επιλύσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ε, ε, διασφαλίσουμε την προστασία ε, ατόμων. Κάθε μορφή υγείας, βίας κατά των γυναικών είναι ε, επίθεση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αποτελεί το θεμέλιο όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται. Στα κράτη-μέλη μας, ωστόσο, υπάρχει έλλειψη ε, κατάλληλης προστασίας για τους πολίτες μας κατά της ε, βίας μεταξύ προσώπων και έχει αποδειχθεί ότι τα κράτη μας έχουν αποτύχει στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι η έμφυλη βία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και το, το γεγονός ότι ο βαθμός της βίας, η ένταση της βίας πολλές φορές ε, παραγνωρίζεται. Χρειάζεται, ε, χρειαζόμαστε μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε την έμφυλη βία. Χρειαζόμαστε εκστρατείες ευαισθητοποίησης στις κοινωνίες μας προκειμένου να αυξήσουμε την βούληση των θυμάτων αλλά και την εμπιστοσύνη τους στις ε, ε, αρμόδιες αρχές προκειμένου να καταγγέλουν ε, τη βία και να χρησιμοποιούν τα μέσα προστασίας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι μόλις 7 τέτοιε εντολέ έχουν εκδοθεί από την προθεσμία ε, εφαρμογής που ήταν τον Ιανουάριο του 2015. Ο αριθμός αυτός αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι πολίτες μας, αλλά ακόμη και οι οργανώσεις που διαστροπιούνται ε, στο θέμα αυτό δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει εντολή προστασίας. Γι' αυτό και χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα η κατάρτιση των δημόσιων αξιωματούχων που εργάζονται επαγγελματικά με τα θύματα όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από κάποιους εμπειρογνώμονες ότι το εργαλείο αυτό είναι δύσκολο στην ε, χρήση του λόγω της περιπλοκότητας ε, και των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των νομοθετικών πλησίων στα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να ισχύει αλλά τίποτα στην μακρά ευρωπαϊκή ιστορία δεν ήταν εύκολο. Μπορού, μπορέσαμε να κατακτήσουμε και να επιτύχουμε πολλά επειδή υπήρχε βούληση. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να μπει στο επίκεντρο της προσοχής μας η ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών μας. Και νομίζω ότι με συνεργασία θα καταφέρουμε να ε, υπερβούμε τα προβλήματα. Πρέπει ε, να τηρήσουμε και να σεβαστούμε τις ε, αρχές ε, που κατοχύρουν στη συνθήκη αλλά και στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Να εξαλειφθεί η βία και να υπενθυμίσουμε ότι το βασικότερο καθήκον μιας κοινωνίας δεν είναι η προστασία των συνόρων ή των θεσμών, αλλά η σωματική ακαιρεότητα και η ελευθερία κάθε πολίτη. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια θα συμπεριλαμβάνει την προσωπική, την ατομική προστασία, προστασία και θα προστατεύει τους πολίτες από την ε, έμφυλη ε, βία. Για να επιτευχθεί όμως ένα τέτοιο σκοπός χρειάζεται αφοσίωση και προσπάθειες από την ε, Επιτροπή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις ε, υποχρεώσεις της. Αυτά ε, από εμένα προς το παρόν. Έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω και τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ, κυρία Ράια Πόστ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Πεσσαρίλη, στην Ευχαριστώ πολύ. και σας Πρόεδρε ευχαριστούμε και την Συμπρόεδρο. Καλώς όρισαν όλοι όσοι βρισκόνται εδώ, όλο μας το κοινό που ενδιαφέρθηκε για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Συμφωνώ 100% με την ε, Σοράγια όσον αφορά το πώς έχουν τα πράγματα με την εντολή. Και για την τιμή στην προηγούμενη θητεία να είμαι η συγγήτρια επί ισπανική προεδρία είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είχαμε πει ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Και τελικά βρέθηκε το καινούργιο εργαλείο προστασία, ώστε να υπάρχει κάποιο μηχανισμό δυναμικό, αποτελεσματικό και να είναι κάτι άσχετο με την γραφειοκρατία και αυτό που το οποίο θέλουμε είναι να αποφύγουμε ένα, ένα, ένα θύμα, ας πούμε ένα θύμα βίας κατά των γυναικών να μπορεί να μετέλθει αυτού του ε, εργαλείου και ε, επίσης θέλαμε εάν το θύμα μετακινηθεί σε άλλη χώρα να μπορεί να καταγγείλει. Όμως θα έπρεπε να παρακάμψει το γλωσσικό πρόβλημα της καταγγελίας στην άλλη χώρα. Και Όλα ε, αυτά τα προβλήματα θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε η ευρωπαϊκή εντολή ε, αντιστοιχούσε σε μια τέτοια προσπάθεια συνεπούς πολιτικής για το θέμα δικαιοσύνης, ελεύθερης και δικαιοσύνης. Δεν είναι θέμα σύγκλησης των εθνικών νομοθεσιών, είναι θέμα δικαστικής συνδρομής. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα ε, με αυτόν το μηχανισμό το 2010 παρουσιάστηκε αυτή η οδηγία η οποία ε, έπρεπε να καλύψει αυτές τις χίλιες γυναίκες οι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτοντας την χώρα τους από κάποια μέσα προστασίας σε σχέση με τη βία που ασκήθη εναντίον τους ε, θεωρήθηκε ότι έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα σωρό γυναίκε που θα μπορούσαν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε όμω, ότι τελικά μόνο 7 τέτοιε εντολέ εξεδόθησαν και μόνο 7, ενώ είχαμε τόσες χιλιάδες συνολικά στις χώρες. Άρα αυτό είναι πλήρης αποτυχία. Επομένως, γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχουμε 1.200 ή 1.200 που ε, χρειάζονται αυτή την διασυνορική προστασία. Αλλά, δυστυχώς, η πρόβλεψή μας ήταν λανθασμένη. Δεν τα πήγαμε καλά όσον αφορά με τις προθέσεις μας. Ο, για διάφορους λόγους απέτυχε αυτή η προσπάθεια, πρώτα όλα σε κάποια κράτη-μέλη. Η βία κατά των γυναικών αντιμετωπίζεται από το ποινικό δικαιο. Αλλού όμως είναι θέμα αστικού δικαίου. Ε, αυτό περίπλεξε τα πράγματα. Ε, επίσης ε, και τα ασφαλιστικά μέτρα προστασίας τα μέτρα απομάκρυνσης όπως τα λέμε διαφέρουν από χώρα σε χώρα άρα οι επαγγελματίες που έπρεπε να, τα, να εφαρμόσουν ε, αυτήν την ε, οδηγία λέγανε ότι είναι δύσκολο ακριβώς επειδή ήταν θέμα αλλού ποινικού, αλλού αστικού δικαίου έτσι μπλέχτηκαν τα πράγματα για την έντολη προστασία και πέραν της δυσκολίας εφαρμογής αυτής με ποινικό αστικό δίκαιο Είχαμε τη ε, μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επεσήμανε ότι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Δεν εξεδόθησαν, είπαμε, αρκετέ οδηγίες. Ε, και έτσι δεν ε, έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ένα κεντρικό αρχείο, μητρό, πρωτόκολλο, άρα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τι γίνεται. Η περιπλοκή επίσης που εμπόδισε την εφαρμογή ε, της οδηγίας ευσκέντρης εργίας αυτό ήταν. Και έτσι είχαν προβλήμα να ωφεληθούν και οι δικαιούχοι. Αυτά τα, τα, τα ευάλωτα πρόσωπα. Επίσης δεν υπήρξε αρκετή ενημέρωση προς τις εθνικές αρχές που έπρεπε να κάνουν την εφαρμογή. Επίσης πρόβλημα συντονισμού, πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Ήταν και θέμα μετάφρασης, πολύ σημαντικό για κάτι που θα χρησιμοποιηθεί διασυνοριακά. Πρέπει όμω να υπάρχει κάτι που να προστατεύει τα θύματα και ακριβώ. Ε, είχα κάνει εγώ την ε, εισήγηση για το πρώτο μα ε, ψήφισμα στην προηγούμενη θητεία και υπάρχει το 2002 αντίστοιχο ψήφισμα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώ θα προχωρήσουν γιατί όλα αυτά αποτελούν ενιαία δέσμη μέτρων. Να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία, να τα συντεριάξουμε για να δούμε πώς μπορούν να προχωρήσουν. Είχαμε τον χάρτη πορείας της Βουδαπέστης για την προστασία των θυμάτων. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που βελτίωσαν τις ρυθμίσεις για τα θύματα. Πρώτα-πρώτα λοιπόν το δικαίωμα του να ακούγεται το θύμα, δικαίωμα συμμετοχή στην ποινική διαδικασία, δικαίωμα στην μετάφραση, στην ε, δικαστική συνδρομή και πολλά άλλα. Δεν καλύπτεται βέβαια εδώ πέρα η εντολή προστασίας. Έτσι θα βαγίστηκαν τα δικαιώματα των θυμάτων. Μπορούν επομένως αυτά να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την εντολή προστασίας. Άρα έτσι μπορούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα στη σημερινή προσπάθεια. Μόνο τέσσερις εντολές, εκτός με στην Ισπανία, δύο στην Γερμανία και μία εντολή προστασία στην Ιταλία πουθενά άλλη εντολή. Ας είμαστε επομένως ειλικρινείς. Είπαμε ότι κρούμε τον κόσμο κινδύνου και από την άλλη μεριά δεν καλύπτονται όλες τις γυναίκες χρειάζονται την εντολή. Γι' αυτό σας λέω ότι μου προξενεί έκπληξη το ότι ενώ υπάρχει τόση ζήτηση κάτι έλειψε, κάτι λείπει στην προσπάθειά μας. Θα πρέπει βέβαια όλα τα κρατημέλη που έχουν προσχωρήσει να εφαρμόσουν τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και θα και την προσωρινή φετινή έκθεση για αυτή την ε, συνθήκη. Πρόκειται έτσι να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης ε, για την βία κατά των γυναικών και έτσι πρόκειται να βελτιωθεί και η ρύθμιση για την εντολή προστασίας. Είπαμε, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική κατάσταση, σε κάθε χώρα καλύπτονται άλλα θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της βίας κατά των γυναικών. Δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί τα πράγματα σχέση με την παλαιότερη οδηγία. Αλλά τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η εντολή προστασίας η ευρωπαϊκή. Το θέμα είναι και πώς θα προχωρήσει η υπόθεση των εντολών προστασίας σε κάθε κράτος μέλος και Σωράγια και εγώ σε αυτή την προσπάθεια υλοποίηση της ιδέας θέλουμε τα πράγματα να βελτιωθούν, θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές, τις δύο συνεισηγήτριες καλύτερα, που επισήμαναν τα προβλήματα με το ΙΠΙΟ και ας περάσουμε τώρα στην ακρόαση. Όπως είπε η κυρία Μπεσερέλ, Ας ακούσουμε τι έχουν να πούν οι εμπειρογνώμονες, ιδίως όσοι έχουν συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αξιολόγηση από πλευράς EPRS. Η κυρία Λάουρα Ρωμάν και ο κύριος ε, Ολιβέρας που θα έχουν το μικρόφωνο στη διάθεσή τους για 20 λεπτά. Σας παρακαλώ να παρουσιάσετε τα συμπεράσματα της μελέτης σας στις δύο επιτροπές. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η Λάουρα Ρομάν και εγώ Εργαζόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Ταραγώνα και αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι η οδηγία του 2011 1999 99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, μια υπόθεση που μας ανατέθηκε και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες ερεύνης του Κοινοβουλίου για αυτή την έρευνα που μας ανατέθηκε και θα τα κάνουμε ως εξής. Ε, εγώ να σας πω δύο λόγια για αυτήν την ε, εντολή προστασίας όπως είπαμε είναι κάτι το περίπλοκο θα προσπαθήσω να σας τα πω όμως απλά και κατόπιν η Λάουρα Ρωμάν πρόκειται να σας παρουσιάσει τα συμπεράσματα του που κατέληξε αυτή η μελέτη και Ακριβώς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έχουμε σε διάφορα κράτη-μέλη την ε, εσωτερική νομοθεσία και εδώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία μέσων προστασίας. Αυτά τα μέσα προστασίας μπορεί να αφορούν το τον ε, ένοχο μπορεί να ε, αφορούν τον εγκλισμό του σε φυλακή, τον, την απομάκρυνσή του, διάφορα μέτρα, διαφορετικές διαδικασίες. Αλλά μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ε, αυτά τα μέτρα πρώτα-πρώτα στην κατηγορία των μέτρων του αστικού δικαίου. Αυτά έχουν σχέση με το κοινωνικό δίκαιο, έχουν σχέση με ε, το διαζύγιο ε, και αυτά τα μέτρα ε, περιλαμβάνουν κάποια μέτρα υποκατάστασης της φυλάκισης ε, ή τέλο πάντων περιοριστικά της ελευθερίας κατόπιν επομένως της, της δίκης. Και επίσης υπάρχουν και κάποιο είδους ασφαλιστικά μέτρα κατεπίδοντος χαρακτήρα που είναι πολύ συγκεκριμένα, κρατούν συγκεκριμένο μικρό διάστημα και έχουν κάποιο διοικητικό χαρακτήρα με την έννοια ότι αυτά όλα προέρχονται από την αστυνομία. Δεν τα δει αστυνομία, υπάρχει μια ε, κρίση, ε, ο ένοχος από το θύμα διαχωρίζονται και λαμβάνονται αυτά τα διοικητικού χαρακτήρα καταπήγοντα μέτρα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας στο, στο περιθώριό της μάλλον γιατί δεν κρατούν πολύ καιρό οπότε επ' αυτής της βάσεως για όλους αυτούς τους διαφορετικούς κανόνες των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προέβη στην θέσπιση ενό συνόλου κανόνων, ώστε όταν χρειάζεται προστασία και έχει προστασία μάλλον κάποιο θύμα, ε, πηγαίνει από το ένα κράτο μέλος σε άλλο. Οπότε θα πρέπει πάλι να ισχύουν αυτά τα μέτρα και τα περισσότερα από τα οποία έχουν σχέση με τη δικαστική συνδρομή. Επομένως, αυτά τα οποία βλέπετε ε, στην διαφάνεια ε, αφορούν ακριβώς αυτήν την αμοιβαία αναγνώριση και αυτή η δικαστική συνεργασία και συνδρομή της αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δικαστικές αρχές διαφορετικών κρατών μελών και ε, η μία αρχή έχει εκδώσει την Ευρωπαϊκή Εντολή η οποία ισχύει για όλο τον κοινό χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Άρα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ιδέα. Ε, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας με αυτή την οδηγία βασικά είναι μηχανισμός δικαστικής συνδρομής και σε δεύτερη φάση είναι μηχανισμός προστασίας αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι για κάθε ότι, ότι, πρόκειται για ε, συνεργασία και προστασία όλα αυτά τα οποία βλέπετε στο slide είναι σχετικά με την αποτελεσματικότητα και υλοποίηση εφαρμογή της οδηγίας. Έχουμε δύο αποφάσεις πλαίσιο οι οποίες έχουν σχέση με κάποια μέτρα εποπτείας ή ελέγχου όπως είπαμε την προσωρινή κράτηση ή ή φόρους αποφυλάκηση. Ε, και επίσης έχουμε και τον κανονισμό 606 603 λεωμιλήτρια του 2013 και επίσης με αυτή την οδηγία έχουμε κάποια εσωτερικά μέτρα ποινικού χαρακτήρα. Και έτσι καταλήγουμε σε την οδηγία για την ε, εντολή προστασία. Αλλά έχουμε και τα μέτρα ε, αστικού δικαίου τα οποία σχετίζονται με τον κανονισμό που βλέπετε εδώ. Όπως είπε η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ, η συγκίτρια, δεν έχουμε τώρα μόνο θέμα δικαστικής συνδρομής, έχουμε και θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων. Έχουμε δηλαδή την οδηγία για τα θύματα και από την άλλη έχουμε την οδηγία για την εντολή προστασίας. Ε, έτσι θεωρούμε ότι το ένα νομοθέτημα μπορεί να καλύψει τα κενά του άλλο. Πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτή η εντολή προστασίας. Για να υπάρξει αυτή η εντολή προστασίας πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εν κινδύνο σε ένα κράτος μέλος. Και αυτό το πρόσωπο πρέπει κάποια δικαστική αρχή ή άλλη αρχή ισοδύναμη αντίστοιχη να το εξασφαλίσει κάποια μέτρα, μέτρα είτε ποινικού είτε αστικού δικαίου. Να αποφασιστεί επομένως από αυτό το πρόσωπο, αυτό το θύμα ε, να θέλει να μεταβεί από το κράτος έκδοσης στο κράτος εκτέλεσης. Ε, τότε συντρέχει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας Είπαμε τα, τα ποινικά φορούν την οδηγία και τα αστικά φορούν τον κανονισμό. Οπότε για να, για να ξαναδούμε το, μάλλον για να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Next. Έτσι εξηγείται η σχέση οδηγίας με τις αποφάσεις πλαίσιο. Εάν το θύμα και ο θήτης, ο ένοχος, αλλάξει κράτος μέλος, τότε δεν ισχύει η οδηγία. Εφαρμόζονται οι αποφάσεις πλαίσιο. Άρα τα ίδια μέτρα, αλλά επί τη βάση της, των οδηγιών πλαίσιο. Για τον ένοχο του εγκλήματος και όχι για το θύμα. Το θύμα έχει την εντολή προστασίας, αλλά εάν ο ένοχος του εγκλήματος αλλάξει και αυτός χώρα, τότε ισχύουν οι οδηγίες πλαίσιο. Εάν επομένως αυτός από το κράτος έκδοσης πάει σε τρίτη χώρα, σε αυτή την περίπτωση, ο ένοχος θα υφίσταται κάποια μέτρα, τα οποία θα γίνονται δυνάμει των αποφάσεων πλαίσιο. Το δε θύμα θα έχει τύχει κάποιας εντολής προστασίας από το κράτος εποπτείας. Είναι περίπλοκο, μα γι' αυτό και το εξηγούμε. Επόμενη διαφάνεια. Αυτά τα μέτρα είπαμε γνωρίζουν μια ποικιλία από κράτος σε κράτος. Όμως, η εντολή προστασίας καλύπτει αυτά τα τρία μέτρα που βλέπετε εδώ. Πρώτα πρώτα, απαγορεύεται κάποιος να έρθει σε επαφή με το θύμα, να πλησιάσει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και να έρθει σε επαφή. Εάν επομένως υπάρχουν κάποια μέτρα του εσωτερικού δικαίου κράτους μέλους δεν αναγνωρίζονται από την εντολή προστασία. Οι βοήθειε, οι ρυθμίσεις σχέση με την οικογένεια δεν αναγνωρίζονται από την εντολή προστασία. Μόνο αυτά καλύπτει η εντολή προστασία που σας ανέφερε. Τώρα για κάποια ε, το τι είδους μέτρα έχουμε. Πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί ο ένοχος. λέμε για τα μέτρα απομάκρυνσης. Είναι αυτά τα μέτρα τα οποία λείπτουν καταρχήν κάθε θύμα αλλά κυρίως αφορούν τη βία κατά των γυναικών ή παρενόχληση. Αυτά τα τρία μέτρα είναι αυτά τα οποία καλύπτονται τόσο από την οδηγία και από τον κανονισμό και στις αποφάσεις πλαίσιο που σας ανέφερα. Αυτά τα τρία μέτρα και όχι άλλα. Επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά την διαδικασία, πώς λειτουργεί η εντολή προστασίας. Όπως σας είπα, για να υπάρχει θα πρέπει πρώτα-πρώτα να έχουμε εσωτερικά μέτρα προστασίας. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή εντολή προστασία σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο και εφαρμόζεται επί τη βάση όσων προβλέπονται στο κράτος έκδοσης και όταν έρχεται η ώρα της εκτέλεσης στο κράτος εκτέλεσης ε, τότε πάλι εφαρμόζεται το εσωτερικό δίκαιο του κράτους έκδοσης άρα πάντοτε όλα αυτά εξαρτώνται από το εσωτερικό δίκαιο. Τώρα το αν υπάρχει αντιστοιχεία από το ένα κράτος στο άλλο αυτό και όχι ταυτό της προστασίας ότι είναι ακριβώς η ίδια από το ένα κράτος στο άλλο δεν χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία το θύμα για άλλη διαδικασία Αρκεί το ότι υπάρχει η εντολή προστασία την οποία και επικαλείται. Εάν τώρα προβλέπετε στο δίκαιο ότι και άλλοι μπορούν να ζητήσουν αυτά τα μέτρα, Τέλος πάντων μόνο το θύμα μπορεί να επικαλεστεί την εντολή προστασία. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να επικαλεστεί το θύμα την εντολή, δεν προβλέπεται δεν προβλέπεται διαδικασία επακροατηρίου. Όμως, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος ε, συνεχίζει να υπάρχει, αν ο κίνδυνος έχει ενταθεί κλπ. Ένα θύμα λοιπόν, μια γυναίκα βρίσκεται σε κάποιο οίκο υποδοχής και προστασίας και έτσι και αυτό είναι μυστικό, δεν ξέρει το, ο ένοχος που θα τη βρει. Και ας πούμε ότι αλλάζει η χώρα πάει για λόγου οικογενειακού στη χώρα προέλευση. Οπότε όμω τότε ο κίνδυνο αυξάνεται. Γιατί αν δεν ξέρει ο ένοχο που βρίσκεται αυτή, όταν αλλάζει κράτο, τότε θα συνθεί με την οικογένειά τη. Οπότε και το, και το θύμα, α πούμε, ότι είναι από την ίδια χώρα. Οπότε οι συγγενεί μπορούν να, να του πούνε, ξέρει, η πρώην, η πρώην σου βρίσκεται εδώ. Οπότε είναι αυτή η περιπτώση αυξάνεται ο κίνδυνος αλλά αυτό μόνο ε, από δικαστές, από δικαστικού μπορεί να ζυγιστεί. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι όταν ε, έχουμε επίκληση εντολής προστασίας θα πρέπει να ξέρουμε ότι άλλαξε χώρα όποτε εκδίδεται τέλος πάντων εντολή προστασίας. διότι τεκμέρεται ότι ο ένοχος ξέρει ότι θα φύγει από τη χώρα το θύμα. Άρα γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε αποτελεσματικοί να υπάρχει ταχύτης. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία, έχουμε τους κανόνες μεταφοράς της οδηγίας στο εστρικό δίκαιο που ορίζουν το πώς γίνεται και με τι προθεσμίες πώς γίνεται αυτή η μεταφορά πώς έχουμε τα εκτελεστικά μέτρα, πώς λαμβάνονται αυτά. Είναι βέβαια και θέμα επιμέλειας των δικαστών, αλλά κυρίως των διοικητικών αρχών. Να είναι ξεκάθαρο που δεν είναι ακόμα με τι διάβλους διαβιβάζονται από το ένα κράτος στο άλλο οι εντολές προστασίας. Όταν λοιπόν έχει γίνει η επίκληση της εντολής προστασίας όλα εξαρτώνται από τη χώρα προέλευσης. Άρα κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ κράτους εκτέλεσης και κράτους έκδοσης. Δεν είναι αυτονόητο όμως ότι υπάρχει τέτοια συνεχής επαφή Βεβαίως και επιβάλλεται να υπάρχει εναρμόνιση όσον αφορά τις κυρώσει για την παραβίαση της εντολής προστασίας. Σε κάθε κράτος μέλος άλλα ορίζει το κάθε ιστορικό δίκαιο. Αλλού προβλέπονται χρηματικές ποινές, αλλού ποινές στερητικές ελευθερίας. Άρα χρειάζεται εναρμόνιση. Εν κατακλείδιο όσον αφορά αυτό που θα σας πω εγώ, οι εντολές προστασίας έχουν τα υπέρ και τα κατά. Όλα εξαρτώνται από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Δεν υπάρχει εναρμόνιση. Δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ του τι ρυθμίζεται σε κάθε κράτος μέλος. Και τώρα να δώσω στην συνάδελφο την ε, σκητάλη για να μας πει τι αποκομίσαμε από τη μελέτη. Καλημέρα σας. Όπως έλεγε η συνάδελφος, ο στόχος αυτής της ε, μελέτης ήταν να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η εντολή προστασίας. Το 17 μας ανατέθηκε αυτή η μελέτη στην αρχή και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο τέλος πάντων. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη είχαμε σαν αφετηρία τη μελέτη των υφισταμένων ρυθμίσεων. Οπότε και γι' αυτό και θέλουμε να δούμε τρία επίπεδα πρωτα Πρώτα-πρώτα τις διατάξεις της οδηγίας, όπως είπε η νέος, και η οδηγία ρυθμίζεται τα της έκδοσης και εκτέλεσης της εντολής προστασίας. Δεύτερον, έπρεπε να δούμε πώς γίνεται η μεταφράση στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα κρατη που το έχουν κάνει και τι έγινε φέτος. Επίσης, κατά τρίτον, έπρεπε να αναλύσουμε τους κανόνες δικαίου κάθε κράτους μέλους, τα μέσα δηλαδή προστασίας που προβλέπουν οι ιστορικές νομοθεσίες. Εδώ ήταν το θέμα, γιατί είπαμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό εδώ είναι η ποικιλία, η πολυμορφία στις ρυθμίσεις. Όλα αυτά κάλυψε αυτή η μελέτη, όλα αυτά τα νομοθετικά ζητήματα στη συνέχεια του Δάφνη που ήταν ένα άλλο παλιότερο project αναλύσαμε όλες τις ε, πληροφορίες προσπαθήσαμε να δούμε τι έχει συμβεί από τον Ιανουάριο του 2015 τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία του τι έγινε μέχρι και σήμερα για να δούμε, να ενημερωθούμε ε, έπρεπε να κάνουμε κάποιο είδου γκάλωπ, κάποιο είδου ερωτηματολόγιο 28 ερωτήματα υπήρχαν που απευθύναμε στις αρχές των κρατών μελών. Οι περισσότερες υπηρεσίες ήταν υπηρεσίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης ή των Υπουργείων που χειρίζονται τα ευρωπαϊκά θέματα. 19 απαντήσεις πήραμε και σε αυτή την πρώτη φάση υπήρχε κάποια δυσκολία γιατί ήρθαμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές αλλά με δυσκολία γιατί δεν έχουμε κάποιο είδους ε, κατάλογο ενιαίο για το ποιες είναι οι αρμόδιες τέτοιες αρχές στην ε, Ένωση. Πού να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε για τις πληροφορίες. Δυσκολία επομένω επαφής με αυτές τις αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πού θα τους βρούμε αυτούς όλους. δυσκολία υπήρχε και από πλευρά των εθνικών αρχών, γιατί δεν υπάρχει πουθενά ούτε σε κράτος μέλος, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιο είδους πρωτόκολλο για τις εκδοθήσεις εντολές προστασίας. πότε γι' αυτό και με επιφύλαξη λάβουμε υπόψη τις 7 εκδοθήσεις εντολές. 7. 7 βρήκαμε Θεωρούμε ότι αυτό έχει προσωρινό χαρακτήρα, γιατί μπορεί κάτι να μας ξέφυγε. Κάπου σε κάποιο κράτος μέλος να υπάρχει κάποια άλλη εντολή. Πάντως, θεωρήσαμε ότι με αυτό το στοιχείο βρισκόμαστε ενώπιον δραματικής καταστάσεως, όπως είπε η συγγήτρια. αυτή τη διετία. Φυσικά και υπάρχουν θύματα τέτοιων εγκλημάτων που άλλαξαν χώρα. Δεν ζήτησαν εντολή προστασία και δεν προστατεύτηκαν από αυτή την ρύθμιση που θα όφιλε να είναι αυτόματη. Το 2010 είπαμε ότι έχουμε 10.000 γυναίκες που προστατεύτηκαν από διάφορα μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2016 στην Ισπανία εκδόθηκαν 9.500 ε, μέτρα προστασίας. 28% αυτών των μέτρων ζητήθηκαν από αλλοδαπές. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα σήμερα έχουμε θύματα τα οποία μετακινούνται από το ένα κράτος στο άλλο και δεν ζητούν ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Οπότε, εν ώψη όλων αυτών των στοιχείων και όσον αφορά τις μελέτες και τα αποτελέσματα που πήραμε για αυτές τις στατιστικές, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά τις εκδοθήσεις εντολές, αλλά και για το μέλλον, το τι μπορεί να προκύψει πρώτα-πρώτα, ότι το βασικό είδος βίας το οποίο σχετίζεται με την εντολή προστασίας είναι η βία κατά των γυναικών στα πλαίσια ενός ζευγαριού, μιας σχέση. και είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε εντολές και σε περίπτωση παρενόχλησης και σε περίπτωση ε, μαστροπίας. Και βασικό μέτρο εδώ είναι ο διαχωρισμός και απομάκρυνση τέλο πάντων του ενόχου από το θύμα της μαστροπίας. Επίσης, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει το στοιχείο το διασυνοριακό. Δηλαδή, όταν το θύμα για λόγου ε, εργασιακούς, για λόγου ε, οικογενειακούς, συνήθως μετακινείται. πολλέ φορές κάθε μέρα από τη μία χώρα σε άλλη, που είναι κοντά η μία στην άλλη. Οπότε η εντολή προστασία μπορεί να εδώ να είναι χρήσιμη και χρειάζεται αναβάθμιση συντονισμού των διαφορετικών κρατών μελών γιατί τα μέσα προστασία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν συνεχώς και στις δύο χώρες μέλη. Τρίτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να επισημάνουμε το ότι σε πολλές εντολές προστασίας εμπλέκονται ανήλικοι. Τα παιδιά που μετακινούνται μαζί με τις μητέρες τους. Η σχετική οδηγία δεν περιέχει διατάξεις όσον αφορά αυτά τα ιδιαίτερως ευάλωτα πρόσωπα. Γιατί εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και τους αναπήρους. Και όπως είπαμε προηγουμένως, όπως τα είπαμε με την συντάκτρια, την εισηγήτρια, έχουμε πει ότι αυτό θα πρέπει να προσεχθεί. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοια πρόσωπα σε κάποια εντολή προστασίας χρειάζεται συμπληρωματική επίκληση τις οδηγίες για τα θύματα. Οπότε έτσι καλύπτονται και αυτοί ιδιαίτερα ευάλωτοι, τα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα. Δεν προβλέπει εντολή προστασία να έχουμε πάνω από ένα πρόσωπο του ίδιου κοινωνικού πυρήνα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μνήμα όταν έχουμε θέμα ανηλίκου. Άρα κοντά στην εντολή για τον γονιό του, τη μητέρα του, να βγαίνει εντολή προστασία για τον ανήλικο. Επίσης είπαμε ότι έχουμε πολλές φορές μετανα... μετακίνηση σε διαδοχικά πάνω από ένα ή δύο δύο κράτη-μέλη. Το θέμα είναι να μονεύεται όμως σε ποιο κράτος θα πάει το θέμα. Έχουμε εδώ λοιπόν στο θέμα εδώ των διαδοχικών εντολών πάνω από ένα κράτος ή να έχουμε ταυτόχρονα εντολές και αυτές να απευθύνονται και να διαβιβάζονται σε πάνω από ένα κράτος μέλος. Άρα εδώ επίσης χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, περισσότερη ενημέρωση των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών. Τέλος, μια το στο μέλλον. Τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Όταν ο κίνδυνος της βίας ή η βία δεν είναι σωματική αλλά γίνεται με άλλα σημερινά μέσα μέσω του facebook, μέσω του ίντερνετ τα σχετικά μέτρα τώρα είναι πιο περίπλοκα τα μέσα προστασίας είπαμε ότι έχουμε μετακίνηση σε κράτος όπου προβλέπεται περισσότερη προστασία. Ε, σε αυτή την περίπτωση, λογικά το θύμα θα είναι δικαιούχος αυτών των έξτρα μέτρων προστασίας καλύτερου επίπεδου. Αλλά οπότε λέμε ότι έχει συμπληρωματική προστασία στο νέο κράτος μέλος. Είναι κάποια, κάποιες παροχές κοινωνικές για αυτά τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων. Τέλος, όταν ο σκοπός της μετακίνησης του θύματος είναι μόνο και μόνο να διαφύγει από τον διώκτη, τον ένοχο, τότε χρειάζεται η εντολή προστασίας ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση τη υποτροπής από πλευρά του ενόχου. τελικό στόχο της εντολή προστασία είναι να υπάρχει ουσιαστική προστασία. Να μην υπάρχει πάμε υποτροπή του εγκλήματο και γι' αυτό χρειάζεται κάποιο είδου εποπτεία, παρακολούθηση του πώς πάνε τα μέτρα προστασίας στο κράτος εκτέλεσης. Τι πρόκειψε από την μελέτη, ότι έχουμε κάποιους ε, αριθμούς, ε, κάποιο τηλέφωνο που μπορεί να πάρει κανείς και αυτό παρέχει κάποια προστασία και αυτό υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη, αυτά τα κατεπήγοντα νούμερα πρώτων βοηθειών ας πούμε. Ε, επίσης υπάρχουν κάποια ε, gadget μπορεί το, κάποιος να φορέσει ένα τέτοιο gadget και να επισημαίνεται που είναι με, με GPS και αυτό αφορά και το θύμα και τον ένοχο. Χρήσιμα αυτά. Όμως υπάρχουν κάποιο είδους προβλήματα όταν αυτά είναι χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού πρώτα-πρώτα κοστίζουν πολύ αυτές οι συσκευές δεύτερον το, το, το, το πεδίο λειτουργίας όταν να καλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές υπάρχουν ασυμβατότητες. Τεχνική ασυμβατότητα. Από το ένα κράτος στο άλλο. Γι' αυτό, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν. Μιλούμε για κάποιες εφαρμογές σε smartphone. Ή υπάρχουν σε κάποια κρατημέλη στα κινητά λοιπόν, με αυτές τις εφαρμογές μπορεί άμεσα να υπάρχει ενημέρωση για τον κίνδυνο. Είναι άμεση, σχεδόν αυτόματη η επαφή με την αστυνομία. Γεωεντοπισμός. Πολύ αποτελεσματικά αυτά τα συστήματα. Επίσης βοηθούν τους ε, αναπήρους αυτές οι εφαρμογές και βοηθούν και σε περίπτωση που κάποιο θύμα δεν γνωρίζει την ε, γλώσσα της χώρας όπου πήγε. Γιατί υπάρχουν ε, εικονίδια, υπάρχουν ε, κάποια βιντεάκια σε νοηματική γλώσσα και όπως είπαμε βίντεο σε περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Άρα είναι πολύ θετική ιδέα η χρήση της τεχνολογίας για να δούμε κατά πόσο πιάνουν τόπο τα μέτρα προστασίας. Πόσο αποτελεσματικά είναι την επόμενη διαφάνεια. Α, εδώ είναι το τελευταίο μέρος της παρουσίασης μας για να σας πούμε για κάποιες ε, ιδέες μας, για κάποιες προτάσεις, κάτι που μας φαίνεται ότι είναι σημαντικά στα οποία πρέπει να σταθούν. Πρώτα-πρώτα, είμαι θα ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση πληροφόρηση του θύματος. Είναι λογικό βέβαια αυτό και να μπορεί να κάνει ε, έτοιμα χορήγηση εντολής το θύμα. Αλλά ακριβώς το θύμα θα πρέπει πρώτα πρώτα να ξέρει, όχι να, να ξέρει ότι πρέπει να ζητήσει την εντολή, αλλά να ξέρει ότι υπάρχει εντολή, ως πώς θα τη ζητήσει. Επίσης, η ενημέρωση για όλη τη διαδρομή της διαδικασίας της εντολής να ξέρει το θύμα σε ποιον θα απευθυνθεί όταν πάει στο κράτος εκτέλεσης, να ξέρει ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές που θα την προστατεύσουν και με τι μηχανισμούς. Να γνωρίζει το θύμα τι θα γίνει σε περίπτωση που ο ένοχος, ο διώκτης την πλησιάσει παρά την εντολή απαγόρευσης προσέγγισης. Να ξέρει το θύμα, το τι δυνατότητες υπάρχουν, τι υπάρχει για να βοηθηθεί στο κράτος εκτέλεσης. Ε, γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, αυτή η ενημέρωση προς το θύμα. από τους επαγγελματίες, από αυτούς που εμπλέκονται, δηλαδή δικηγόρους, υπαλλήλους Υπουργείου Δικαιοσύνης, αστυνομικούς, κοινωνικές, επικοινωνικούς λειτουργούς, όλοι, όλοι οι φορείς και οργανώσεις που βοηθούν τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων να ληφθεί υπόψη επομένω οι περιπλοκότες, οι φραγμοί σε αυτό το μέτρο και άρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση του θύματος στην δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Να διευκολύνουν και να υπάρχει επίσης νομική αρρωγή, να υπάρχει ε, εξασφάλιση συνηγόρου. Να ακούγονται τα θύματα. Να μπορούν να εξηγήσουν τα πραγματικά περιστατικά και έτσι να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που περνά το θύμα. Και βέβαια να φροντίσουμε για την άρση των γλωσσικών φραγμών. Δωρεάν να υπάρχει ερμηνεία και μετάφραση σε σχέση με τη συνεννόηση του θύματος, των θυμάτων τέλο πάντων, με τις αρμόδιες αρχές. Πριν βάλουμε τελεία να σας πούμε ο, για την εντολή προστασία ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν είναι γνωστό. Ούτε καν από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάντε σεμινάρια, κάντε εκστρατείες ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες του κλάδου. Για αυτούς που πλαισιώνουν την εντολή προστασίας και βέβαια χρειάζεται συντονισμός κρατών μελών, συντονισμός των διαφόρων υπηρεσιών. Άρα χρειάζεται να υπάρξει κάποια κεντρική υπηρεσία και να επισημαίνεται, να είναι γνωστό ποιε είναι οι Να υπάρχει κάποιο είδου μητρό, αρχείο, πρωτόκολλο και σε επίπεδο ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρωμάν, κυρία Ολιβάρε, για την παρουσίαση του θέματος η κυρία Λουσία Αβέλες, δικαστής και εκπρόσωπος του Ισπανικού Συνδέσμου Γυναικών Δικαστών, που είναι και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών Δικαστών. Όμως θα τα πει σε βίντεο και λόγω τεχνικών πτυχών, λόγω του μήκους και της ταχύτητας ε, η διερμηνία θα σας δώσει μια σύνοψη και όχι μια πλήρη μετάφραση. Χαίρετε. Καλή σας μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα για το έργο που κάνετε για την Ευρωπαϊκή Διαταγή προστασίας. Είμαι Ισπανίδα, ζω στην Καταλωνία. Η πολιτική κατάσταση κάνει κάπως δύσκολο να λάβω απόφαση να εγκαταλείψω την χώρα έστω και για λίγες ώρες. Θα κάνω λίγα σχόλια. για την έννοια που έχουμε, για τις έννοιες που χρησιμοποιούμε στην Ισπανία δηλαδή, για την βία μεταξύ των δύο φίλων. Όταν ο σύντροφος μιας γυναίκας ή ο σύζυγος προβαίνει σε βίες ενέργειες εναντίον της. Και όσα από αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διαταγής Προστασίας. Ναι. Έχουμε σχετική νομοθεσία στην Ισπανία. που περιλαμβάνει και την έννοια της βίας μεταξύ των φίλων και τη σχετική προστασία. Τα συζητούμε αυτά στην Ισπανία εδώ και καιρό. Και έχουμε αρχίσει ήδη από το 1995, όπου πρώτο άρχισε να χρησιμοποιείται η έννοια της βίας μεταξύ των φίλων για να μεταφράσουμε το gender-based violence που λένε στα αγγλικά. Το 2004 αρχίσαμε να, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ως κοινωνία το βάρος των βιών αυτών πράξεων. Μόλις λοιπόν πριν από 13 χρόνια συνειδητοποιήθηκε στην Ισπανική κοινωνία η βαρύτητα αυτής της βίας. Για την ώρα έχουμε βέβαια την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την Istanbul Convention, που περιγράφει τις έννοιες αυτές για όλα τα είδη βίας κατά γυναικών. Τις σχετικές έννοιες περιλαμβάνει η νομοθεσία μας, για συμπεριφορές δηλαδή ιδιαίτερης βίας, όπως αναγκαστική γάμη, οικονομική βία, ακροτηριασμός των γυναικείων ε, ε, αναπαραγωγικών οργάνων, εμπορία, σωματεμπορία σε βάρος γυναικών, για γενετήσια εκμετάλλευση, σεξουαλική παρενόχληση και ούτω καθεξής. Υπάρχει και αριθμός γυναικών που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα νούμερα. μεταξύ 1968 και 2010 μετρούμε 829 θύματα. Πρόκειται για τρομοκρατία μεταξύ φίλων που έχει στοιχίσει και τη ζωή παραπάνω από χιλίων γυναικών μεταξύ 2003 και 2017. Και αυτά είναι τα επίσημα νούμερα. Τα, τα ανεπίσημα νούμερα είναι ακόμα υψηλότερα. Το 2017 μόνο έχουν ε, δολοφονηθεί 39 γυναίκες. Οχτώ ε, από αυτές είχαν ζητήσει και είχαν λάβει ευρωπαϊκή διαταγή προστασίας και όμως τελικώς δολοφονήθηκαν. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα επίσημα νούμερα και αναφέρονται σε φόνους από την πλευρά δηλαδή που δράστες ήταν οι σύζυγοι κάθετος σύντροφοι των γυναικών αυτών. Το 2015 που έγινε σχετική έρευνα από την Ισπανική κυβέρνηση έδειξε επίσης σημαντικά νούμερα για γυναίκες άνω των 16 ετών που ένα 10,7% από αυτές είχαν υποστεί βία, είτε κτυπήματα, είτε απόπειρα στραγγαλισμού και ούτω καθεξής. Από συντρόφους συζύγους ή πρώην συντρόφους συζύγους. Παρ' όλα αυτά έχουν μειωθεί οι καταγγελίες τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαταγές προστασίας. Χρειάζεται μια ενεργός προσέγγιση από τον δικαστή ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. «5.300 περίπου έχουν ε, χορηγηθεί διαταγές προστασίας Τα λέω αυτά και σας λέω και τα νούμερα για να εξηγήσω ποια είναι η διάσταση του προβλήματος όχι μόνο της ποια είναι οι διαστάσεις της βίας μεταξύ των φίλων Το πιο σημαντικό είναι αυτή η αίσθηση έλλειψης προστασίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είτε από τις αστυνομικές αρχές είτε από τις δικαστικές. Και καλούνται οι γυναίκες να εξηγήσουν γιατί έχουν περάσει χρόνια σιωπής.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 entrando de lleno los τώρα ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ε, όταν έρχεται η ώρα της ιοξιολόγησης γιατί έχουν δοθεί τόσο λίγες εντολές προστασίας. Δεν υπάρχουν πάντοτε οι προϋποθέσεις ούτε ώστε να εκδοθεί μια εντολή και οι στρατηγικές σε περίπτωση κάποιων ε, τουριστών που έχουν υποστεί αυτή την βία, οι γυναίκες δεν ε, καταγγέλουν τα όσα έχουν υποστεί γιατί δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη, κρίσιμη μάλλον και σημαντική η στάση της αστυνομίας. Ε, και πολλές φορές υπάρχει και πρόβλημα γλωσσικό γιατί βρίσκονται στη χώρα για πολύ λίγο διάστημα κάποιοι ως τουρίστες. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Είναι εδώ να υπάρχει αυτόματη έκδοση της ε, εντολής είτε από δικαστική είτε από εισαγγελική αρχή. Το πρόβλημα αυτό το ξεπερνάμε έχοντας ε, αξιόλογες πλήρε πληροφορίες και ενημέρωση. Αυτό δεν γίνεται πολλές φορές και άρα ε, έχουμε πολλές φορές την έκδοση μιας εντολής εθνικής ισπανικής εντολής προστασίας και τελικά ζητείται όμως ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και θα πρέπει σε 72 ώρες να γίνει α, ακρόαση από το δικαστή, αλλά ένα διαφορετικό δικαστή που δεν ξέρει καλά το φάκελο, τη δικογραφία. Οπότε θα πρέπει να αξιολογήσει ο δικαστής πληροφορίες από το θύμα ειδικό για την περίοδο της προστασίας. Αλλά θα πρέπει να ξέρει τις αρχικές ε, να έχει τις κατάθεση και να βρει τα αποδεικτικά στοιχεία. Δύσκολο αυτό γιατί συνήθως γίνεται συνοπτική διαδικασία όσον αφορά ε, αυτά τα εγκλήματα της βίας κατά των γυναικών. Πολλές φορές υποτιμάται ο κίνδυνος από τη βία. Πολλές φορές οι Ισπανοί δικαστές δεν ενεργούν ως Ευρωπαίοι δικαστές, δεν έχουν την εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμως προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στην συμφωνία του 11 της Κωνσταντινούπολης, ε, στην οποία προσχώρησε πανή το 14. Όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν από κάποιο είδου νομικά μέσα, τα οποία προβλέπονται ακριβώ για βία κατά των γυναικών, αλλά χρειαζόμαστε δικαστικού και αστυνομικού ειδικά εκπαιδευμένου. Υπάρχει μια επιτροπή, το ΟΗΕ, που μελετά το θέμα της καταπολέμησης πάσης δυσμενούς διακρίσεως κατά των γυναικών και έχει διαβιβάσει στην Ισπανία διάφορες συστάσεις όπως το να υπάρχει κάποιο είδους ε, εύλογη αποζημίωση προ τα θύματα, να εξεταστεί ε, το σε ποιε περιπτώσει οι γυναίκε δεν έχουν επαρκή προστασία και ε, να ρυθμιστούν και τα θέματα των ανηλίκων, τα δικαιώματα των ανηλίκων, να ακούγονται οι ανήλικοι, τα παιδιά, πάρα πολύ σημαντικά αυτές αποφάσεις θα πρέπει να υποχρεωτικά να εκπαιδεύονται οι δικαστές στα θέματα οικιακής βίας και να αναγνωριστεί το ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι στην Ισπανία και ο φόρτος εργασίας των δικαστών. Ο πρόεδρος Μωράης, ε, με συγχωρείτε που κάπως άκομψα διακόπτω την προβολή του βίντεο. Ε, ευχαριστούμε πολύ την δικαστή ε, για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση, αλλά έχουμε πίεση χρόνου Δυστυχώ, έχουμε ψηφοφορία στι 11, έχουμε λοιπόν κάποια πίεση χρόνου και έχουμε και ακόμη έναν ομιλητή. Και κάποια στιγμή χάθηκε και η μετάφραση για κάποια λεπτά. Ευχαριστούμε πάντως την δικαστή για την παρέμβασή της. Πολύ πιθανόν όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο μπορούν ε, να, μπορούμε να το διαθέσουμε και μπορούμε ενδεχομένω να δώσουμε και κάποια μετάφραση, γραπτή δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο για να παρακολουθήσουμε την ε, προβολή, γιατί έχω και ε, μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο. Προχωρούμε στον επόμενο ομιλητή μας, εκτελεστικό διευθυντή του Victim Support Europe, Θέλετε να λάβετε το λόγο. Α, εσείς, είναι η κυρία Μπεσερέλ, γιατί είναι υποχρεωμένη να αποχωρήσει. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί θα χρειαστεί πιθανότατα να φύγω πριν από το τέλος της συνεδρίασης γιατί το χρονοδιάγραμμα ε, είναι λίγο πιεστικό. Θέλω να ευχαριστήσω όλες σας. Πολύ σημαντικό, όπως είπατε, η μαρτυρία αυτή πολύ σημαντική και θα είναι χρήσιμη για μας για να τις συνεισηγήτρες δηλαδή, για να τις συζητήσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα είμαστε σε επαφή και βέβαια και θα ε, λάβω υπόψη και την παρέμβαση του ε, εκτελεστικού διευθυντού. Ευχαριστώ. Ελπίζω η Σοράγια, η ετέρα των συνεισηγητριών, να μπορέσει να παραμείνει κοντά μας μέχρι τέλους. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο πραγματογνώμονα και μετά θα δώσουμε τον λόγο στα μέλη. Ο κύριος Λέβεντ Άουταν, εκτελικός διευθυντής του Victim Support Europe. Δέκα λεπτά μην τα υπερβείτε κύριε ε, Διευθυντά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ερωτήσεις μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καθώς και εσάς κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ για την ευγενή σας πρόκληση, πρόσκληση Είμαι διευθυντής του Victim Support Europe. Είμαστε δηλαδή ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών, οργανώσεων που στηρίζουν τα θύματα ε, και στηρίζουμε περίπου 2 εκατομμύρια θύματα ανά έτος. Ε, είμαι ενώπιόν σας και διότι έχω εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν είχε γίνει η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασίας. Έχω λοιπόν κάποιο σχετικό ιστορικό εκεί δεν δούλεψα πάνω στις EPO από τότε, στην εφαρμογή δηλαδή των Ευρωπαϊκών Διαταγών Προστασίας. Είναι σημαντικό βέβαια αυτό να το ε, συζητήσουμε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, στις ερευνήτριες για το έργο τους, το οποίο μου θύμισε πολλά από τα ζητήματα που συζητούσαμε τότε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι ενδιαφέρον που ακούσαμε τα προβλήματα και τα ενδεχόμενα προβλήματα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο, ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί τον κίνδυνο μπορεί εν τέλει να εντοπίσει το θύμα ξανά και ξανά και ακόμη και αν έχει αλλάξει ε, τόπο διαμονής ή κατοικίας. Είναι ε, ενδιαφέροντα και θεμελιώδη θέματα αυτά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για μένα πάντως θα ήθελα μάλλον να το προσεγγίσω από διαφορετική διάσταση. Το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι η ζήτηση για Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασία. Η ερώτηση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν χιλιάδε χιλιάδων γυναικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο που, ε, κινδυνεύουν και χρειάζονται προστασία. Αναμφίβολα είναι μείζον, πολύ μείζον το πρόβλημα. Υπάρχει όμω και ένα ξεχωριστό ερώτημα. Υπάρχει πράγματι ζήτηση από την πλευρά των θυμάτων για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασία. Γνωρίζω δεν υπάρχουν στατιστικέ. Όμω οι καταγγελίε προέρχονται ας αφήσουμε την ΙΠΙΟ ε, ζητούν προστασία όταν φεύγουν στην Αλοδαπή οι οργανώσεις το ζητούν γιατί ζητούν όλο περισσότεροι άνθρωποι και οργανώσεις προστασία εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τις οργανώσεις μας για τις προτεραιότητες, για την ανάπτυξη μια στρατηγική, Έχουμε ένα τετραετές πρόγραμμα που έχουμε εγκρίνει τώρα. Μιλούμε για εθνική προστασία κυρίω. Πρώτη ερώτηση μου λοιπόν είναι αυτή. Ποιο, πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Έχω σημειώσει εδώ ορισμένε ερωτήσεις που είναι σχετικές με αυτό. Πόσοι... Πόσοι άνθρωποι... Ποιο είναι το πρόβλημα, πόσοι άνθρωποι γίνονται θύματα όταν φεύγουν στο εξωτερικό. Ακούσαμε βέβαια κάποια παραδείγματα, αλλά πού βρισκόμαστε, γιατί αυτά θα μας δείξουν ποιος είναι ο πληθυσμός που καλούμαστε να προστατεύσουμε. Πόσοι ζητούν όταν φεύγουν στο εξωτερικό την προστασία και δεν τη λαμβάνουν. Και αν τη λάβουν γιατί τη λαμβάνουν αργά. Πόσοι άνθρωποι έλαβαν προστασία στο εξωτερικό αλλά δεν ήταν επαρκής. Ακούσαμε την δικαστή να μιλά για οκτώ περιπτώσεις όπου δόθηκε η Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασίας και όμως τελικώς δολοφονήθηκαν οι γυναίκες. Άρα δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα στο εξωτερικό, οι γυναίκες αυτές πέφτουν θύματα στο εξωτερικό. Ποια είναι η προστασία που προσφέρει το μέτρο, γιατί αυτό θα μας δείξει και εάν λειτουργούν όντως τα εθνικά μέτρα ή όχι και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να προστατεύσουμε τις γυναίκες αυτές στην πράξη. Πόσα άτομα που έχουν ε, εθνική προστασία, ε, εθνική ε, Διαταγή προστασίας θέλουν να φύγουν πόσοι αισθάνονται ασφαλεί, αισθάνονται ασφαλεί για να φύγουν. Και πόσοι άνθρωποι, λέει πάντοτε ο μιλητή, χρειάζονται ή θέλουν ευρωπαϊκή διαταγή προστασία, αλλά αποθαρρύνονται. Ποιε είναι οι περιστάσει για τη, για τη μετακίνησή του, πώ λειτουργεί η διαδικασία. Τα σκέπτονται οι άνθρωποι αυτά όταν φεύγουν στο εξωτερικό. Πόσα χρόνια μετά από τη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή προστασίας σκέπτονται να φύγουν στο εξωτερικό και κατά πόσο επηρεάζει η εμπειρία εκείνη. Ας δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι πιο χρήσιμες δράσεις για να προστατευτούν οι γυναίκες. Μιλούμε για 100.000 διαταγές προστασίας τον χρόνο. Περίπου 40.000 από αυτές προέρχονται μόνο από την Ισπανία. και 95% πάντως από ένα μικρό αριθμό χωρών. Αυτό ήδη λέει κάτι για το πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί είναι τόσο δραστήρια η Ισπανία και άλλες χώρες όχι. Δεν νομίζω ότι, εκεί, ότι στην Ισπανία υπάρχει περισσότερη οικιακή βία από ό,τι αλλού, έστω και αν υπάρχουν βέβαια ε, παραλλαγές. Και τι γίνεται με τις ΕΠΟ που έχουν εκδοθεί. Τι γίνεται με τις ΕΠΟ αυτές. Γιατί μόνο 7 ΕΠΟ Ποιε είναι οι περιστάσει που οδήγησαν στην εκδοσία αυτών και από αυτέ τι 7, 4 είναι πάλι μόνο από την Ισπανία. Γιατί τα θύματα αυτά ζήτησαν την υπηόπια ή ήταν τα χαρακτηριστικά τη προσωπική του περίπτωση, ε, πώ ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα τη ΕΠΙΟ. Ποια ήταν η εμπειρία του από την διαδικασία υποβολή αίτηση, από την ανταπόκριση των αρμοδίων. Πόσο κράτησε η διαδικασία. Υπάρχει ικανοποίηση τα θύματα όντως προστατεύθηκαν. Θεωρούν δηλαδή ότι όντως λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή ε, Διαταγή Προστασίας. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν στην αρχή, γιατί πολλά από τα άλλα ερωτήματα είναι περισσότερο ε, εικασίες. Δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα που ε, μπορούν να προκύψουν από την έκδοση της, της διαταγής προστασίας. Σημαντικό λοιπόν να δούμε και τι γίνεται όταν ζητούν και δεν εκδίδεται. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα θύματα στο εθνικό επίπεδο και διασυνοριακά. Εγώ δεν λέω ότι η διαταγή προστασία, η ευρωπαϊκή δηλαδή, δεν είναι αναγκαία, αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία που να μα δείχνει αν είναι αναγκαία, πότε είναι αναγκαία. Έχουμε λοιπόν, ξαναλέω, χιλιάδε ανθρώπων, γυναίκε, οι οποίε γίνονται θύματα οικιακή βία κάθε χρόνο και πρέπει πράγματι να δράσουμε και να δράσουμε αποφασιστικά. Και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό που είναι η σύμβαση της Ισταμπούλ, της ε, Κωνσταντινούπολης που προβλέπει δράση για την προστασία των γυναικών. Χρειάζεται να γνωρίζουμε λοιπόν ποιες είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες μέσα στον μηχανισμό αυτό. Ποιες είναι οι σημαντικότερες δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα ποιε είναι οι επιπτώσει που είναι τα προβλήματα, που μπορεί να προσφέρει η προστιθέμενη αξία η Ευρώπη. Αν τα εξετάσετε αυτά, γυναίκες που μπαίνουν σε καταχρηστικές σχέσεις, πώς μπορούν να ξεφύγουν από τις καταχρηστικές σχέσεις οι γυναίκες, με ποια προστασία, με ποια προετοιμασία, με ποια βοήθεια μακροπρόθεσμα, πώς μπορούμε να διώξουμε τους παραβάτες, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, ερώτημα είναι Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Χρειάζονται πρακτικά μέτρα για να προωθηθούν όλε αυτέ οι δράσει. Και πώ εφαρμόζεται το άρθρο 18 τη Οδηγία για την Προσέγγιση των Θυμάτων, που λέει όταν είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν και διαδικασίε του εθνικού δικαίου για την σωματική προστασία των θυμάτων και των οικογενειών του. Εδώ ανοίγει ένα παράθυρο για εθνική δράση. Ακούμε τι παρεμβάσει αυτέ σήμερα και ορισμένε από τι παρεμβάσει αυτέ αναφέρονται τα προβλήματα στο εθνικό επίπεδο με την λειτουργία των εθνικών διαταγών προστασίας. Αν αυτές οι εθνικές διαταγές προστασίας δεν αποδίδουν, τότε η ΕΠΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν υπάρξει καν η αίτηση ή η ζήτηση. Δύο προτεραιότητες. Πρώτο, αποτελεσματική ενημέρωση των θυμάτων, εντός και εκτός δικαιικού συστήματος συστήματος μάλλον απονομής δικαιοσύνης. Αυτό θα τις βοηθήσει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν οι διαταγές προστασίας και τι πρέπει να κάνουν για να τις αποκτήσουν τις διαταγές προστασίας. Και τα μέτρα των εθνικών συστημάτων πρέπει να εξεταστούν για να δούμε αν λειτουργούν σωστά. Αυτό σημαίνει να υπάρχουν, να προβλέπονται σωστά μέτρα τα οποία να είναι εύκαμπτα, να βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Εδώ πράγματι η Ισπανία είναι πρωτοπόρος αποτελεσματικότητα των διαταγών προστασίας. Δεν αρκεί να πεις «Α, δεν επιτρέπεται να πλησιάσει την γυναίκα α ή β». Χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την προστασία για όταν πρόκειται να συμβεί το κακό. Τα μέτρα αυτά μπορούν να εγκριθούν σύντομα. Υπάρχουν οι αναγκαίες προστασίες. Έχουμε το παράδειγμα όπου η αστυνομία τα, βλέπει, τα προβλέπει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία. Γιατί υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, φόνων γυναικών οι οποίες περίμεναν ακόμα να δραστηριοποιηθεί ο δικαστής. Προβλέπεται εκπαίδευση σε αστυνομικές αρχές, εισαγγελικέ αρχές, δικαστές για να αντιδρούν. Αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που δρούν επιτόπου την ανάγκη να δράσουν άμεσα. Ακούμε ξανά και ξανά για την πρακτική ότι ε, δεν χρησιμοποιείται, ότι οι γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ε, ζητήσουν τη λήψη των μέτρων αυτών λόγω πολιτιστικών αιτίων κλπ. Χρειάζονται αποτελεσματικές πρακτικές προστασίας, αποτελεσματικές τεχνολογίες. Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Και όσον αφορά την οδηγία προστασίας θυμάτων, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προηγούμενο και έχει δώσει την ευκαιρία να γίνει δουλειά πάνω σε αυτά τα πρότυπα γιατί κατά τη γνώμη μου η οδηγία εγκρίθηκε και προτάθηκε κυρίως στην βάση της εμπιστοσύνης. Το άρθρο 82 παράγραφος 2 μιλεί για δικαστική συνεργασία. Χρειαζόμαστε μέτρα δικαστικής συνεργασίας. Όμως το θεμελιώδες εδώ είναι όταν υπάρχει έλλειψη δικαιωμάτων μέτρων πρέπει υπέρ των θυμάτων. Πρέπει οι δικαστές, οι αγγελίε, οι αστυνομικοί κτλ. να μπορούν να βασίζονται, να έχουν μια εμπιστοσύνη στην λήψη των μέτρων. Αν υπάρχουν μέτρα τα οποία προστατεύουν τα θύματα της οικίακή βίας και εναντί άλλων κινδύνων, μπορούμε να έχουμε πραγματικά γνήσια εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών και των ανθρώπων που ε, ασχολούνται με τα θέματα αυτά, των practitioners, πολλές ερωτήσεις, αλλά ότι καλύπτουν ορισμένα από τα θεμελιώδη θέματα που ανοίγονται εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ορισμένες ερωτήσεις για τα όσα είπατε, αλλά προτιμώ να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, αν θέλουν είτε να παρέμβουν είτε να ερωτήσουν. Και στο τέλος θα σας ζητήσω να συνοψίσετε. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω ποιος θέλει να παρέμβει για δύο λεπτά. Στέτινα. Ευχαριστώ. Φυσικά, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες διότι αυτά που είπατε ήταν πολύ σημαντικά για εμένα. Στη ζωή μου πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ζήσει ποτέ από κοντά έμφυλη βία, παρά μόνο στον Οθέλο. Νομίζω ότι μου ανοίξατε τα μάτια δηλαδή. Και τώρα έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα για το πόσο τρομακτική και αποκρουστική είναι η έμφυλη βία. Ακούστηκε πολύ συχνά αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός 7 είναι γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης χρήσης ε, αυτής της εντολής προστασίας αποτελεί δείκτη ε, ότι υπάρχει ανάγκη κάτι να αλλάξει. Και εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Έχουμε αυτήν την εξαιρετική μελέτη που εκπονήθηκε. Γενικώ όμως υπάρχει μία καταφανής έλλειψη πληροφοριών θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τη δική σας γνώμη. Τι πιστεύετε ότι θα είναι πιο σημαντικό στο μέλλον. Να αναθεωρηθεί, να αναδιατυπωθεί η οδηγία περί Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας ή θα ήταν καλύτερο να, να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ δικαστικών λειτουργών, την ευαισθητοποίηση στα, ε, για τα θύματα. Ευχαριστώ κύριε Στατίνα Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος στις ε, εισηγήτρες θα ήθελα να δώσω το λόγο στο τέλος. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ ως μέλος. Εγώ ήμουν ενεργό μέλος αυτής της Επιτροπής όταν ε, υποβλήθηκε αρχικός η σχετική πρόταση και είχαμε συζητήσει τότε κάποια θέματα που έθεσε και ο κ. Άουταν αλλά και κάποια άλλα ζητήματα που τέθηκαν από άλλους συναδέλφους. Οι χώρες που είχαν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν ε, και που την επέλεξαν αυτή τη δυνατότητα πρέπει πλέον να πάρουν απόφαση να, ε, να ε, συμμετάσχουν. Υπήρχε τότε εκείνη την περίοδο ανάγκη να να, να δημιουργηθεί, να θεσπιστεί αυτή η εντολή προστασίας. Αυτή η δυσανάλογη χρήση από ένα ή δύο κράτη ενδέχεται να καταδεικνύει και μια έλλειψη όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και είναι πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτό το εργαλείο που θα μπορούσε να είχε αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό ως μέσο προστασίας είτε συμπληρωματικά προς τα εθνικά μέτρα είτε και με σκοπό τη βελτίωση του εθνικού πλαισίου λήψης μέτρων. Και γι' αυτό θα ήθελα από αυτό το βήμα να επισημάνω κι εγώ ότι η φάση της εφαρμογής ήταν απογοητευτική. Ε, πράγματι φαίνεται ε, να έχει ξεχαστεί το εργαλείο αυτό. Σε αντίθεση με την πολύ πρώτη περίοδο μετά την θέση σε εφαρμογή της ε, εντολής προστασίας, όπου φαινόταν ότι υπήρχε, ε, υπήρχε ε, γνώση και που πολλές χώρες επέλεξαν τελικά να συμμετάσχουν. Ποτέ βεβαίως η εντολή προστασία δεν θεωρήθηκε ότι θα ήταν πανάκια και ότι θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα. Ε, πάντοτε είχε ένα χαρακτήρα συμπληρωματικό ε, που αφορούσε ιδίως τις διασυνοριακές υποθέσεις. Αλλά είναι ακριβώς αυτές οι υποθέσεις όπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Αυτά. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Προτού ξαναδώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Η Κομισιόν ακούω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ήταν σφάλμα δικό μου. Δεν υπήρχε στα, στα, στις σημειώσεις μου ε, ότι θέλει να παρέμβει και η Κομισιόν με συγχωρείτε ήταν, ε, ήταν σφάλμα δικό μου Τοποθέτησα από την Κομισιόν παρακαλώ έχετε το λόγο συγγνώμη δεν, έχω, δεν ξέρω ούτε το όνομά σας παρακαλώ συστηθείτε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ιζαμπέλ Περινιό, τμήματάρχης ε, ε, σε ζητήματα ποινικού δικαίου Και πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε το θέμα αυτό με μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συζήτηση που έγινε σήμερα και για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Η σωστή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και η εφαρμογή του κανονισμού για την ε, αμοιβαία αναγνώριση σε δικαστικές υποθέσεις, σε αστικές υποθέσεις είναι ε, ύψης της προτεραιότητας για την Κομισιόν. Όλα τα κράτη-μέλη που δεσμεύονται από την οδηγία EPO έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα μέτρα μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και γι' αυτό ε, ε, ε, χρειάστηκε ε, αρκετός χρόνος έως ότου ε, λάβουμε όλες τις ε, πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο σημαντική προτεραιότητα τώρα για εμάς είναι να ετοιμάσουμε την έκθεση την οποία θα παρουσιάσουμε ε, του χρόνου. Συμμεριζόμαστε και εμείς την απογοήτευση που εκφράσατε και λυπόμαστε και εμείς που το μέσο αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί ε, επαρκώς. Οι εξηγήσει που ακούστηκαν από τον κύριο Λεφαλτό είναι σε έναν βαθμό ε, και δικές μας εκτιμήσεις. Ε, διότι είμαστε και εμείς σε επαφή με τα κράτη-μέλη για να μάθουμε για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείται αρκετά αυτό το μέσο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, κοινοποιήσει κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές που έχουν συστήσει και όλα αυτά μας βοηθούν για να δούμε πώς μπορεί να προωθηθεί αυτό το μέσο. Το έχουμε βάλει στο, στην πύλη e-justice, στην ιστοσελίδα του, του δικτύου ε, δικαστικής συνεργασίας και στο δίκτυο δικαστικής κατάρτισης όπου στο εκπαιδευτικό υλικό έχει πλέον ενταχθεί και ειδική εκπαίδευση για τις δικαστικές αρχές γύρω από την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, ώστε, όπως ακούσαμε και για την περίπτωση της Ισπανίας, να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί ε, έχουν γνώση ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να ερευνούμε το ζήτημα, ε, να καταβάλουμε προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση σε όλους τους τομείς ε, που άπτονται των δικαιωμάτων των θυμάτων. Επίσης, ε, ε, δίνουμε και ε, χορηγίες και επιδοτήσεις μέσω διαφόρων προγραμμάτων της, στον τομέα της δικαιοσύνης. Καταβάλουμε προσπάθειες λοιπόν για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη-μέλη και στις 29 Ιανουαρίου του 2019 θα διοργανώσουμε και ένα ειδικό εργαστήριο ε, με θέμα την, ε, τα δικαιώματα των θυμάτων. Θα γίνει εκεί μια συζήτηση με πυρογνώμους από τα κράτη-μέλη σε μια πλειάδα θεμάτων. Μεταξύ αυτών θα είναι και η βία κατά των γενικών και η εφαρμογή των εντολών προστασίας. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη δική μας πλευρά κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί πραγματικά είναι σοκαριστική η κατάσταση που επικρατεί σε κάποιες χώρες, ιδίως στην Ισπανία, αλλά όχι μόνο στην Ισπανία. Η κατάσταση αυτή αφορά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι και το βασικό, λέει ο Πρόεδρος, ε, ότι η κατάσταση αυτή αφορά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει ε, είναι ε, η φάση της εφαρμογής και ακριβώς να γίνει η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας ένα εργαλείο που θα αξιοποιείται και ότι θα ε, το γνωρίζουν τουλάχιστον οι αρχές στα κράτη-μέλη. Έστω και ως συμπλήρωμα προς τα εθνικά μέτρα που ενδεχομένως να λαμβάνουν. Ευχαριστώ πάντως. Ε, βρισκόμαστε προς το τέλος ε, της ακρόασης μας. Μπορώ να σας πω επίσης ότι θα σας διαβιβάσουμε τα έγγραφα και τις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε σήμερα. Ξέρετε επίσης ότι η ε, η συνεδρίασή μας αυτή ε, μεταδόθηκε και στο διαδίκτυο, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και θα μείνει και στον σερβερ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πάντως ε, και τα έγγραφα που μας αποστήλατε και που μας παρουσιάσατε θα διαβαστούν στα μέλη των επιτροπών μας. Να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή εντολή προστασία είναι ένα θέμα στο οποίο υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μα, ατομικών ελευθεριών και γυναικών. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στην εισηγήτρια μα, Σωράγια Πόστ, ώστε να κάνει κάποιε καταληκτικέ παρατηρήσει, να συνοψίσει ενδεχομένω τη συζήτηση τα όσα ακούστηκαν σήμερα και να κλείσουμε με εκείνη την σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ, Κλοντ και ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες, τις παρεμβάσεις, τις οποίες βρήκα πολύ σημαντικές για εμάς ως εισηγήτριες. Και είχε πει και η Τερέζα πριν αποχωρήσει ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές. Αλλά και οι πληροφορίες που λάβαμε μόλις από την Κομισιόν είναι πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη, εγώ και η Τερέζα, να ξανασυναντηθούμε με την Κομισιόν για να λάβουμε λεπτομερώς όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, θέσατε πολλά ερωτήματα, κύριε Λεβάντ, και τα, οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βεβαίως θα μας απασχολήσουν και θα είναι πολύ σημαντικά κατά τη φάση σύνταξη της ε, έκθεσής μας. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά, πρέπει να γίνουν γρήγορα, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την εξασφάλιση, για την ασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και νομίζω ότι και η Κομισιόν πρέπει να αποδείξει την, ε, το γεγονός ότι είναι αφοσιωμένη στην σωστή λειτουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Εντολής ε, Προστασίας και χαίρομαι που είχατε αυτή τη φορά τουλάχιστον να μοιραστείτε ε, κάποια θετικά νέα. Πρέπει η Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασία σε παραβάση ε, ε κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και επίσης η Κομισιόν πρέπει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων όπως και αυτή περιγράφεται στην οδηγία. Πρέπει λοιπόν να, ε, γίνουν ε, εκστρατείες ε, ευαισθητοποίησης, έρευνες όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και η Κομισιόν οφείλει να εξασφαλίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των, του, κάθε κράτους μέλους με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Επίσης, πρέπει η Κομισιόν να προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή ε, προτάσεων για την ε, καλύτερη λειτουργία του EPO. Επίσης, πρέπει να δημοσιευθεί ένας κατάλογος των αρμόδιων αρχών ε, σε κάθε κράτος μέλος, των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση ε, των Ευρωπαϊκών Εντολών Προστασίας, για, για, την, ε, για τη διαβίβαση αυτών των εντολών προστασίας, αλλά και των οργανώσεων που υποστηρίζουν και βοηθούν τα θύματα και που ορισμένες φορές διαμεσολαβούν. Επίσης πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, καταγγείλουν ε, την, ε, διαπροσωπική, την βία μεταξύ προσώπων. Η Ισπανία δικαστής αναφέρθηκε πράγματι σε έμφυλη τρομοκρατία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο όρος. Δεν είναι δυνατόν να υποτιμάται ε, ο βαθμός στον οποίο υποφέρουν τα, θέ, τα θύματα, ούτε τα θύματα ε, να ε, ε παρουσιάζονται ως θύτες ε, των ε, αξιόπινων πράξεων των οποίων έχουν υπάρξει θύματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες Ευχαριστήσω όλα τα μέλη των δύο επιτροπών μας για την παρουσία τους εδώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μωράης. Τώρα, 11 η ώρα. 11 η ώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Το λέω αυτό για τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών.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 Σοφή Λιμπαλά, του να σύγχρονα, ασύλληλα. Mr. Chairman, can we get on with this? Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Yeah, I was just waiting for you to say that. Ναι, περίμενα ότι θα το λέγατε αυτό. Γι' αυτό και χτύπησα το σφυράκι μου. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πάσα που μου δίνετε. Παρακαλώ, ας καθίσουμε όλοι. The complicated Everyone have their... Είναι περίπλοκες ε, οι ψηφοφορίες μας. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Έχει... Υπάρχει κάποιος που δεν έχει την κάρτα του μαζί. Ας μας το πει τώρα, όχι αργότερα σας παρακαλώ. Άρα έχετε όλοι τις κάρτες σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Επομένω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι και οι συντονιστέ. όλοι έτοιμοι. Okay, the first vote is on... Πρώτη ψηφοφορία. Κανονισμός 45 του 2001, αναθεώρηση αυτού. Κορνέλια Έρνστ είναι η συγγήτρια. Θέλει το λόγο η συγγήτρια. Αν όχι, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη ψηφοφορία. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας και δεν το λέω τυπικά. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 17. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is still open while people sit down. Ψηφίζουμε ακόμη μέχρι να καθίσουν όλοι. Παρακαλώ καθίστε. I'm just hold on. I'm just giving one or two members some leeway as they sit down. Περιμένω μέχρι να καθίσουν ένα-δυο μέλη τη επιτροπή μα ακόμα τα τελευταία. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε πρέπει να προχωρήσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ε, για το άρθρο 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Okay, colleagues, pause for a moment. The S&D have one... Στους σοσιαλιστές υπάρχει ένας, ένα μέλος που περισσεύει. Λύστε το παρακαλώ αυτό το πρόβλημα. Τέλεια. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 253. Άρχιτη ψηφοφορία. Amendment 253. 253. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε ακόμη. Ψηφίστε ο κύριος Φως δεν βρίσκει την τροπολογία. Με ενημερώνουν, είναι η τροπολογία 253 στην τρίτη σελίδα. Τα ξαναλέω. Ψηφίζουμε επί της 253 που βρίσκεται στη σελίδα 3. Πέρασε της Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 3. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. This is block. closed εγκρίνεται. Τις 112, 13 και 14 θα τις ψηφίσουμε μαζί, 115 και 116 επίσης. Ψηφίζουμε από κοινού. got it? The vote is closed. Εντάξει, τα βρήκατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is Εγκρίνεται. 117. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. That is carried. Sorry, this one we need to come back. We need to. Εγκρίνεται. Okay. Because it was fully adopted, but it was not adopted. Okay. And colleagues, just. Συνάδελφοι, πρέπει να ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 20 γιούρι, την οποία και ξεχάσαμε. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 20 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. The vote is still open. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας συνάδελφος από το ΕΛΚ παραπάνω. Ας βγάλει κάποιος συνάδελφος από το ΕΛΚ την κάρτα του από το μηχάνημα. Παραμένει το πρόβλημα. Παρακαλώ, κάποιος από το ΕΛΚ ας βγάλει την κάρτα του. Ευχαριστούμε. Πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Άρχεται η ψηφοφορία. That's amendment 118. 118. Τροπολογία 118. The vote is closed. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στη συμβαστική τροπολογία του άρθρου 9. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 126. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας. Ο εισηγητής ήταν κατά. Καταψηφίστηκε. Ε, τροπολογία 24. Άρχεται ψηφοφορία. Amendment 24. The vote is open. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 24. Ε, Technical problem. Α, έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι μέχρι να το λύσουμε. Okay. Colleagues, we have to pause. We have a technical problem with the machine. Just pause for one moment. We are on Amendment 24. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να λύσουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα και θα ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 24.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 Okay, colleagues, um, we don't... Συνάδελφοι, ακούστε με σας παρακαλώ προσεκτικά. Συγγνώμη κυρία Ένσχα την δική σας έκθεση. Θα το λύσουμε. Τι έχει συμβεί. Υπήρξε υπερφόρτωση του μηχανήματος. Διότι καταγράφει ότι υπάρχουν 62 παρόντα μέλη που ψηφίζουν. Ενώ μπορεί, μπορούν μόνο 60 μέλη να ψηφίζουν. Τόσα αντέχει το μηχάνημα. Ξεπεράσαμε τα όρια του, του μηχανήματος. Τι θα κάνουμε τώρα. Κύριε Μέλο, παρακαλώ μην αγγίζετε το μηχάνημα. Ακούστε με προσεκτικά. Συνάδελφοι, ακούστε με. Δεν αφορά το ΕΛΚ Θέλω οι συντονιστές να ελέγξουν τον αριθμό των παρόντων μελών τους. Σας παρακαλώ κάτι λίγη ησυχία να σας πω. Κάθε συντονιστής ας ελέγξει τον αριθμό των ε, μελών της πολιτικής του ομάδας που παρίστανται. Θα, θα κάνουμε αυτή την καταμέτρηση και μετά θα ξανακάνουμε έναν έλεγχο. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή και μετά θα... θα προχωρήσουμε κανονικά με την ε, κανονική διαδικασία. Λοιπόν, οι 15, ΕΛΚ. Παρακαλώ ελέγξτε λίγο τον αριθμό των παρόντων μελών σας. Everybody makes a, a vote, a vote like this, in, okay. just to check that. We do a test now, yeah. Okay, I'm presuming from all the hilarity that every... Υποθέτω από τα γέλια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους συντονιστές. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα έναν έλεγχο να δούμε τι θα μας πει το μηχάνημα. Ψηφίστε παρακαλώ, ας κάνουμε μια δοκιμα... Ε, δοκιμή. Ε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Δοκιμαστική ψηφοφορία είναι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε 61 ευρωβουλευτές. Δεν το αντέχει ούτε αυτό το μηχάνημα. Θέλουμε 60. Κάποια ομάδα έχει έναν παραπάνω. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή. Ποια ομάδα έχει έναν ευρωβουλευτή περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να είχε. Uh, Συνάδελφοι, 30 δευτερόλεπτα χρειαζόμαστε και θα το λύσουμε το πρόβλημα. Um, Συνάδελφοι, θα κάνουμε άλλη μία δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν φτάνουμε στον αριθμό 60. Ψηφίστε παρακαλώ, καθίστε και ψηφίστε ό,τι θέλετε για να δούμε πόσοι είναι οι παριστάμενοι. Ξεκινάει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία.

Ωραία, συνάδελφοι, το λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να ξαναπάμε στην ε, τροπολογία 125. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άξιλ, σταμάτα σε παρακαλώ να μιλά. 1, 2, 5. Τροπολογία 125. Άρχιτη ψηφοφορία. Vote is open. The vote is closed. Εγκρίνεται. Τροπολογία 126. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Άρχιτη ψηφοφορία. Vote Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 11. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Vote Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 130. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 132. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 133 και τροπολογία 25 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ. Closed. Η ολοκληρώθηκε. Εγκρίνονται. 134. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Carried. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 31. Άρχιτη ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογίες 39, 41, 43, 44, 45, 46. Από κοινού άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 157. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Amendment 163. Vote open. Τροπολογία 163. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 164. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 165. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 166-167 ταυτίζονται. Ψηφίζουμε από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 42. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 172. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 44. Ψηφίστε παρακαλώ. Σοβαρή ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 177. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 178. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 180. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 182. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 48. Ξεκινά η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 186. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Uh, Συνάδελφοι, κάναμε ένα σφάλμα. Πρέπει να περάσουμε, να επιστρέψουμε στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 184. Δεύτερο τμήμα, να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 184. Βρίσκεται στη σελίδα 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Επανερχόμαστε στην τροπολογία 184 για να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της. Το καταλάβατε όλοι. Το ακούσατε όλοι. Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Ψηφίστε παρακαλώ. Πράσινο κουμπί. Το λέω για το ΕΛΚ. Έτσι, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Σας βοηθάω. We're some tidying up because it's very distracting. Και ο κύριος Βος παρακαλώ να σταματήσει να καταψηφίζει τις δικές του τροπολογίες. Κατα... Ε, απορρίφθηκε, λοιπόν. Πάμε τώρα στην τροπολογία 206. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 53 και 44 που ταυτίζονται Ψηφίζουμε τώρα. Closed. Ψηφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 208 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δεν θα κάνουμε ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 209. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 210. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίφθηκε 212 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 213 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίφθηκε 214 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίφθηκε. 216. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 217. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 219. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 57-220 ταυτίζονται, ψηφίζουμε από κοινού. Τώρα. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 221. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 61. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 226. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 2.51 έως 2.57. Θα τις ψηφίσουμε από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Vote closed. Πέρας εγκρίνονται. Τροπολογία 234, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορριφθήκε. 2.35, 2.36, 2.37 ψηφίζονται από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. σοφορίας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. 238-239 ταυτίζονται. Ψηφίζουμε από κοινού. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση οφορίας Απορρίφθηκαν. Ψηφίζουμε. 240 και 241. 240-241. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote closed. Πέρας. Απορρίπτονται. Okay. Okay. Okay. Yeah.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 Εντάξει, ας προχωρήσουμε. Θα καταγραφεί η ψήφο σας ως αρνητική. 240-241. Ε, Θα καταγραφεί γραπτός ως αρνητική η ψήφο σας. Εντάξει. 242. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη 218. Συγγνώμη. Ψηφίζουμε τώρα επί της τροπολογίας 218 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρασε. Τροπολογία 242. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 243. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε επίσης. 2 ε, η τροπολογία 47 της Επιτροπής Γιούρι. Άρχεται ψηφοφορία. <coughs> Πέραση ψηφοφορίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας από το ΕΛΚ που περισσεύει. Παρακαλώ, ας βγάλει κάποιος την κάρτα του. Πρέπει να επαναλάβουμε τη ψηφοφορία για την τροπολογία 40. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. 244. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 246. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 248. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.50. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Carried. Amendment 255. What is open? Εγκρίνεται. 255. Άρχεται η ψηφοφορια πέρασε. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-48 ταυτίζονται. Ψηφίζουμε από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. Τηλογικέ αναφορέ. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχιτη ψηφοφορία. Συνεχίζουμε να ψηφίζουμε. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 72. Ε, ε, Άρχεται ψηφοφορία. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Συνεχίζουμε να ψηφίζουμε. Τι συμβαίνει. Just check. Is the vote still open? Yeah. The vote is still open. Συνεχίζουμε να ψηφίζουμε στο μεταξύ. Ψηφίζουμε πάντα. Πέρασε τις Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 72. Πέρασε. Κλείστε σας παρακαλώ την ψηφοφορία. Kept it open because I couldn't vote, Ναι, είναι ανοιχτή γιατί δεν μπορούσα να ψηφίσω εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Rejected. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 5, Επιτροπή Γιούρι. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Ψηφίζουμε. Τέλος της Απορρίφθηκε. Τροπολογία 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 76. Ψηφίστε παρακαλώ για τροπολογία 76. πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Ψηφίζουμε. Πέρας, απορρίφθηκε. Τροπολογία 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. Τροπολογίες 5, 7 ταυτίζονται, ψηφίζουμε από κοινού τώρα. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνονται. Τροπολογίε 6 και 8 που επίση ταυτίζονται. Ψηφίζουμε από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας εγκρίνονται. Τροπολογία 7. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 85. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 86. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 13. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 92. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 93. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της Επιτροπής Γιούρη. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και 15. Τροπολογία 15 της Επιτροπής Γιούρη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 97. Άρχεται τη ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται και τελική ε, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση όπως τροποποιήθηκε το κείμενο ψηφίζουμε τώρα ψηφίστε παρακαλώ The vote is closed. ψηφοφορίας 45 υπέρ, 7 κατά, 6 αποχές εγκρίνεται. Και τώρα για την ψηφοφορία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με απόλυτη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 υπέρ, 7 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Ένστ, την εισηγήτριά μας. ο, πρόεδρος κ. Μωράης. Ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε ως τώρα. Έρχομαι στην επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο αποφάσεως του Συμβουλίου για μέτρα ελέγχου για τα ναρκωτικά εισηγητής κύριος Μπόνι. Μία ψηφοφορία. Είστε όλες και όλοι έτοιμοι. Αρχίζει. Με ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ονομαστική μάλιστα. Πέρας. Εγκρίνεται 54 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Κύριε Μπόνι, με συγχωρείτε. Θα έπρεπε να είχε ρωτήσει πρώτα εάν θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι, νεύει αποφατικά. Συγχαρητήρια πάντως κύριε Μπόνι. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η ουσία κύριε Έγκελ, αλλά μου φαίνεται ότι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να είναι. Τρίτη ψηφοφορία, ας κρατήσουμε το ρυθμό, γιατί γνωρίζω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Ας περάσουμε αμέσως στην επόμενη. Η συγητής Μάλιν Μπιόρκ. Σας παρακαλώ κάνετε κάπως ησυχία, ας, προχωρήσουμε σύντομα. Πρόκειται για σχέδιο εκθέσεως για πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο για την μετεκατάσταση Μάλιν Μπιόρκ. Εκπίπτουν ορισμένα πράγματα λόγω της 17 ε, συμβιβαστική. Θα έπρεπε να λέει compromise 17 και ένα άλλο νούμερο. Ελπίζω ότι είναι σαφές όμως η αρχή του κειμένου δηλαδή. Θα ρωτήσω πρώτα, Μάλιν επιθυμείτε να λάβετε το λόγο πριν αρχίσουμε. Σας παρακαλώ σύντομα. Θα είμαι συντομότατη. Ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλες και όλους που είναι παρόντες στην αίθουσα για τη συνεργασία τους, βεβαίως τους και οδησυγητές, όλους τους φορείς, από κυβερνήσεις μέχρι μη κρατικούς οργανισμούς που ε, συνεργάστηκαν. Πρόκειται για τη μοναδική πρόταση που αντικείμενο έχει τους νόμιμους ασφαλείς διάβλους για τη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ. Όλοι χρειαστήκαμε, χρειάστηκε μάλλον να κάνουμε συμβιβασμούς. Ελπίζω τελικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θέση του Κοινοβουλίου που να μας κάνουν υπερήφανε. Ευχαριστώ βεβαίως ε, τη συνεργάτη δέσμου Αμαντίν και άλλες καθώς και τη Γραμματεία και βεβαίως και τους συνεργάτες των άλλων Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ Μαρίν. Να προχωρήσουμε αμέσως. Τροπολογία 117. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 118. Οκ, συμβαστική διακοπές ε, από κάτω. Συμβαστική 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ρωτά ο πρόεδρο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την συμβαστική 1. Όχι, πέρα τη ψηφοφορία λοιπόν, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τρία Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 4 αρχίζει. Κανονικά είναι η σελίδα 6 της λίστας ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Συμβαστική 4. Τέλος, εγκρίνεται και αυτή. Προχωρώ στην συμβαστική 5. <laughs> Βεβαίως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος, ψηφίσατε όλοι, θα παραρωτήσω πρώτα. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 5α αρχίζει η ψηφοφορία. 5α συμβαστική. Ψηφίσατε. Σελίδα 14. 5α. Πέρας. Εγκρίνεται. Όλα βαίνουν καλώς. Παρακολουθείτε όλοι. Ωραία. Συμβαστική 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. 6. Συμβαστική 6. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Συμβαστική 6 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8, σελίδα 19. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 11. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 12 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Συμβαστική τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Είναι η 13 επί του άρθρου 12. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 για το άρθρο 13. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. 1-1-0. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 534. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 18, τροπολογία 115. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 546. Αρχίζει η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος Μωράης. Η 545 πρώτα. 545. Πέρασε. εγκρίνεται αυτή. Τώρα η 546 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 116 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 548. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. Ε, μάλλον 131, με συγχωρείτε. 131. Αρχίζει η φοβορία Πέρας. απερίφθη 132 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 155 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απερίφθη 172 αρχίζει Πέρας. Απορρίπτεται. 225. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 226. 226. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. «237, τέλος, απερίφθη. 247, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. 248, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. Θέλετε να λάβετε το λόγο πριν από την τελική ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχουμε ε- ένα πρόβλημα για την ψηφοφορία. Παρακαλώ να κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα για να μπορούσα να συζητήσω με τους σκιώδες ηγητές της έκθεσης. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ. αδελφή, um, λέει ο Πρόεδρος. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Λίγη υπομονή. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Just have some patience for a minute, but please make it quick. Could the shadows convene very quickly, please? Να είναι γρήγοροι στη συνεννόηση και οι σκιώδεις ηγητές, παρακαλώ. Πριν την τελική ψηφορία. Προβλέπετε το διάλειμμα. Κομμονή λοιπόν. Colleagues, just be patient for another minute. Δείξτε λίγη υπομονή για ένα λεπτό ακόμη. Είναι νομοθετικό έργο και επιτρέπεται η δράση αυτή των εισηγητών. Just be patient for another minute. Thank you. Okay, colleagues, uh, you can resume your seat. Μπορείτε να επανέλθετε στα καθίσματά σας. Παρακαλώ, σύντομα. Πιο κομπ, Κυρίε um, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε πάλι. Έχουμε ένα, μια απόφαση υπό την ισχύ του κανονισμού να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Μπορείτε να με επιτρέψετε να τελειώσω τη φάση μου. Μπορούμε να ψηφίσουμε ξανά ένα άρθρο. Μπορείτε απαιτεί Πριν αρχίσετε να απορρίπτετε τα όσα λέω, επιτρέψτε μου να τελειώσω τη φράση μου. Απαιτεί πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής για να επιτραπεί η κίνηση αυτή. Εάν η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής επιτρέπει, θα επαναλάβω την ψηφοφορία. Ρωτώ λοιπόν, αν υπάρχει πλειοψηφία του συνόλου της Επιτροπής για να επαναληφθεί η ψηφοφορία του 5α επί του άρθρου 5, κάτι το οποίο επιτρέπει ο κανονισμός. Δείξτε παρακαλώ την ε, βούλησή σας με ανάταση της χειρός. Σας παρακαλώ προσέξτε. Ποιοι επιθυμούν να επαναληφθεί η ψηφοφορία του 5α, επί του άρθρου 5. Παρακαλώ να σηκώσει το χέρι ως ναι. Και θα μετρήσουμε τα χέρια. με το χέρι. Αν θέλετε επαλήθευση μπορούμε να κάνουμε και ηλεκτρονικά. Προτιμάτε ηλεκτρονικά. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν να επαναληφθεί ψηφοφορία ψηφίστε ναι με ε, ηλεκτρονικό τρόπο. για το 5. Ψηφίστε ναι τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Πεν, ε, 40, 40 ψήφοι υπέρ είναι σαφές. Ψήφι κατά. Είναι σαφές όμως ότι οι πρώτοι αποτελούν την πλειοψηφία. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν υπέρ της επανάληψης της ψηφοφορίας για την συμβαστική 5α επί του άρθρου 5. Θα επαναληφθεί λοιπόν η ψηφοφορία επ' αυτού του άρθρου. Προσέξτε παρακαλώ γιατί θα κάνουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ κάποια ησυχία. Παρακαλώ να πάυσετε τους διαλόγους. Κάνουμε επα, επανάληψη της ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 5α, επί του άρθρου 5. Η ψηφοφορία αρχίζει. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί η επανάληψη. Άρα ψηφίστε σωστά από την αρχή, όπως επιθυμείτε. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Απορρίπτεται με ψήφους 51 κατά, 8 υπέρ και καμιά αποχή. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Ως συνέπεια της ψηφοφορίας που μόλις κάνατε πρέπει να ψηφιστούν οι 360 και 366. 362, 362 αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ οι συντονιστές να δείξουν πώς επιθυμούν να ψηφιστεί. Για να είναι σαφές αντιλαμβάνομαι ότι συνομιλείτε μεταξύ σας, αλλά για να είναι σαφές, ως συνέπεια της ψηφοφορίας που κάνατε πριν, πρέπει να ψηφιστούν οι 362 και 366. 362 αρχίζει η ψηφοφορία. Ξανά αρχίζει η ψηφοφορία 362. Και σύντομα αν είναι δυνατό. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία 362. Θα κλείσω τώρα. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Απορρίπτεται. 55 ψήφοι κατά, 2 υπέρ. Τώρα, η επόμενη, 366, αρχίζει πάλι η ψηφοφορία. Οι συντονιστές ε, δείχνουν. Πέρας. Απορρίπτεται. 58 κατά, καμία υπέρ. Καλώς. Προχωρούμε τώρα στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 ψήφοι υπέρ, 20 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ψηφίζουμε τώρα. Κύριε Έγγελ, μην εγκαταλείπετε την αίθουσα. Ψηφίζουμε την εντολή. Διαπραγματευτική εντολή. Καθίστε παρακαλώ. Σύντομη ψηφοφορία. Βάλτε πάλι τις κάρτες σας στις σχισμές. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει, όπως είπα, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ 14 κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Thank Σας ευχαριστώ. Έληξε εδώ ο χρόνος ψηφοφορίας.